this is yours, the symbol of the power. Proszę Państwa, otwieramy wspólne posiedzenie. Χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, άρχεται η κοινή συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Με ιδιαίτερη χαρά ήρθαμε εδώ στην αίθουσα αυτή, αφού συνεδριάσαμε από πλευράς μας σε άλλη αίθουσα, Επιτροπή Γεωργίας και ζητήσαμε θέματα γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου και υποδεχτήκαμε αντιπροσωπεία του Υπουργείου Γεωργίας της Βραζιλίας και βουλευτές επίσης και γερουσιαστές καθώς και τον Υπουργό. Πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία και ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση εξ αυτού του λόγου. ...22 γλώσσες έχουμε ε, διερμηνία και τα έγγραφα είναι ηλεκτρονικά στη διάθεσή σας ε, στο e-meeting. Η συνεδρίασή μας επίσης μεταδίδεται απευθείας ε, στο διαδίκτυο. Ε, έγκριση της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών της συνεδρίας 23 Φεβρουαρίου 2015. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίας θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν θέλω τώρα να βγάλω λόγο εδώ, δεν έχω να σας πω άλλα, άλλες ανακοινώσεις. Ο εισηγητής γνωρίζει πολύ περισσότερα και οι διάφοροι εισηγητές από μένα. Η κυρία Μόρη έχει ένα πρόβλημα με τα αεροπλάνα της, με την ανταπόκριση δεν μπόρεσε ακόμα να φτάσει στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε την κυρία Ζώμα να μας παρουσιάσει όλο το θέμα. Και της δίνω μέσω στο λόγο. Παρακαλώ. Για να περάσουμε αμέσως στην ουσία των θεμάτων που μας απασχολούν. Παρακαλώ, δεν θα κάνω άλλη εισαγωγή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα θα συζητήσουμε για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την κλωνοποίηση. Το γνωρίζετε το θέμα. Με εξέπληξε λίγο, φίλο να ομολογήσω, ότι παρόλο που υπάρχει μεγάλη σύμβια μεταξύ των πολιτικών ομάδων και συμφωνία, ήταν πολλές οι τροπολογίες 136. Να το πω ότι υπήρξε φαντασία και δημιουργικότητα. Μπορεί να ακούγονται πολλές, αλλά άμα τις ε, μελετήσει κανείς θα διαπιστώσει ότι και στις τροπολογίες σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούμε και αυτό αντανακλάται. Διότι πολλές τροπολογίες επιζητούν το ίδιο ακριβώς που λέει και το σχέδιο της έκθεσης της συναδέλφου ε, Ζούλια Μόη και της ε, δικής μου ταπεινότητος. Πολλέ τοπολογίε είναι ταυτόχρονα ή πάρα πολύ παρόμοιε μετά όσοι είναι ταυτόσιμε ή πάρα πολύ παρομοιε με τα όσα εμείς είχαμε προτείνει. Για παράδειγμα, το αίτημα ή η απέτηση να απαγορεύεται η εισαγωγή και η εμπορία κλωνοποιημένων ζώων και όλων των ε, ε, απογόνων τους καθώς επίσης και των προϊόντων τους. Επίσης ένα αίτημα ε, να υπάρχουν πιστοποιητικά εισαγωγή για να είναι δεδομένη η χνηλασιμότητα. Το λέει και αυτό το σχέδιο. Επίσης αθλητικές και πολιτιστικές ε, διοργανώσεις να ε, ξερούνται. Αλλά αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος, αυτή η πρόταση. Θέλουμε εξαιρέσεις μόνο για ερευνητικές δραστηριότητες και το προτείνουμε και οι πράσινοι το έχουν προτείνει σε τροπολογία και εγώ με τους συναδέλφους Ντες και Κέστιγκερ έχω κάνει νέα τροπολογία ακριβώς για το θέμα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Ε, Γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν καλύπτεται έπαρκος αυτό, διότι η επικεφαλίδα κάνει λόγο για κλωνοποίηση ζώων που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και αναπαράγονται. Θέλω να εξασφαλίσω ότι ζώα που χρησιμοποιούνται για πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο και αθλητικές ή εκτρέφονται για αυτό το σκοπό ε, καλύπτονται και δεν ε, υπάρχει εξαίρεση από το γενικό κανόνα, από τη γενική απαγόρευση, ότι είμαστε γενικά κατά της κλωνοποίησης. Υπάρχουν τώρα και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις από πλευράς πρασίνων για νέους ορισμούς της και την νεκροποίηση εμβρίων. Βεβαίω υπάρχουν και τροπολογίες ε, που πηγαίνουν προς άλλη κατεύθυνση ε, από το σχέδιο έκθεσης που θέλουν να περιορίσουν ε, τη γενική απαγόρευση μόνο για τα ζώα και τα έμβρια και θέλουν να εξαιρέσουν τους απογόνους και υπάρχουν και άλλες ιδέες που είναι, πηγαίνουν πολύ μακριά, για μένα είναι υπερβολικές, διότι αυτά είναι ανέφικτα πράγματα. Απαγόρευση εισαγωγή για όλα ε, τα προϊόντα από χώρε όπου ε, γίνεται κλωνοποίηση. Ε, αυτό παραπάει, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Ούτε είναι και στόχος μας ε, στο σχέδιο έκθεσης. Λοιπόν, μελέτησα πολύ τις τροπολογίες μαζί με τη συνάδελφο Τζούλια Μόη. Θα το συζητήσουμε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και για τις τροπολογίες. Ε, να δούμε ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε. Και θα παρακαλούσα τώρα τους συναδέλφους να μου εξηγήσουν τις τροπολογίες. Και Νομίζω ότι θέλετε να μας πείσετε για τις τροπολογίες και τη συνάδελφο που απουσιάζει και εμένα ότι έχει νόημα λοιπόν να ακούσουμε τι λέτε για τις τροπολογίες για να τις αξιολογήσουμε θετικά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, προτείνω να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία όσοι ήθιστε να ακούσουμε πρώτα τους ε, σκιώδεις εισηγητές, βεβαίως δεν είναι υποχρεωμένοι, εφόσον θέλουν να μιλήσουν. Έχω εδώ το κατάλογο και μετά θα αναλάβει την Προεδρία ο κύριος Λαβία. Πρώτη κυρία Γιούζο. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα υπερβώ τα δύο λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες μου και Ζόμερ για την έκθεσή τους, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι άκρος πολύπλοκο. Βλέποντας έτσι τις τροπολογίες, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πούμε ότι οι εκθέσεις ε, της ΕΦΣΑ δεν είναι επιστημονικές. Είναι επιστημονικές γιατί συντάσσονται από επιστήμονες και βασίζονται σε επιστημονικά πονήματα, τα οποία έχουν ε, δημοσιευτεί σε επιθεωρήσεις σε επιστημονικές που μπορείς διαβάσουν όλοι. Να μην λέμε λοιπόν ότι γίνεται από έναν απλό υπάλληλο, γίνεται η έκθεση από έναν ειδικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες πάλι, να πω κάτι που λέει ότι είναι κατά της βιοποικιλότητας. Ναι, ισχύει, αλλά το ίδιο ισχύει και για την τεχνητή γονιμοποίηση. Η κλωνοποίηση ενός ζώου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά ε, για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Είναι μια τεχνική βελτίωσης. Επομένως δεν είναι... Αν μετά παραδείγματο για να παραγωγείται από τη γύρια και τα λοιπά είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για την κλωνοποίηση, ένα ζώο δηλαδή το οποίο κλωνοποιείται. Και να μη λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα και τα οποία μάλιστα πλήττουν ε, και την αξιοπιστία του Κοινοβούλου και την ε, σοβαρότητα των επιτροπών μας. Είναι αυτά τα θέματα που θέλω να αναφέρω. Κατά τα λοιπά μπορούμε να είμαστε κατά, ότι είναι κατά τη ε, ευημερία ευεξία των ζώων, ότι δεν θέλουμε κλωνοποίηση. Να το πούμε αν θέλουμε να το πούμε, αλλά μην χρησιμοποιούμε επιχειρήματα που δεν είναι επιστημονικά και που δεν είναι 100% έγκυρα. Αυτά είχα να πω και τίποτε παραπάνω. Ευχαριστώ. Είδατε δεν ξεπέρασα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα κυρία Σάρμπου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα ε, καταρχάς να αναφερθώ στο πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Πολλές τροπολογίες και μεταξύ αυτών και τροπολογίες των συν εισηγητριών μιλούν για το πεδίο εφαρμογής και αναφέρονται σε απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων καθώς και τα ζωικά προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Είναι λογικό. Τα, ε, οι απογονοί είναι μέρος μιας διαδικασίας. Φέρνουν γονίδια που με τρόπο εσκεμμένο, απομονώθηκαν και έχουν αντιγραφεί. Αν είμαστε λοιπόν κατά της κλωνοποίησης θα πρέπει να είμαστε και κατά της αγοράς προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα. Αλλιώς θα δημιουργήσουμε ζήτηση. Εγώ έχω κάνει τροπολογίες για να διευκρινιστεί αυτό. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα ζώα ή τα προϊόντα από τα ζώα αυτά δεν είναι κλωνοποιημένα ζώα ή από ε, απογόνους τους. Έτσι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και οι έμποροι δεν θα ε, πρέπει να ε, ψάχνουν οι ίδιοι τα συστήματα ρεχνηλασιμότητας από που προέρχονται τα προϊόντα αυτά. Γιατί αυτό θα τους επιβαρύνει ιδιαίτερα διοικητικά. Σε ό,τι αφορά τις προσωρινές ή μόνιμες απαγορεύσεις, πολλές τροπολογίες ε, θέλουν φιλοδοξούν να επιβάλλουν μια μόνιμη απαγόρευση και όχι προσωρινή. Συμφωνώ, διότι προσωρινή απαγόρευση θα έδινε ένα μήνυμα πώς να το πω, όχι αρκετά στεναρό. Η τροποποίηση της νομοθεσίας είναι κάτι ε, που ζητείται από κάποιες άλλες τροπολογίες για να λαμβάνουν υπόψη την αίσθηση της κοινή γνώμης. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το λάβει υπόψη ε, γιατί μπορεί να αλλάξει θέση ε, και η κοινή γνώμη ως προς την κλωνοποίηση ή τα τρόφιμα. Και τέλος όλες οι βολιδοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν θέλει ο κόσμος αυτά τα προϊόντα. Και συμφωνώ κι εγώ. Και ως εκπρόσωποι των πολιτών θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή τη θέση και να την ε, εντάξουμε και στην έκθεσή μας αλλά και στις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Η κυρία Αγγιλέρα για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς συμφωνώ και εγώ με τα συγχαρητήρια προς τις δύο εισηγήτριες και την κυρία Σόμερεν προκειμένου που είναι παρούσα. Θα ήθελα να πω το εξής. Οι δικές μου τροπολογίες βαίνουν προς μια κατεύθυνση και μια θέση ίσως ενδιάμεση ανάμεσα στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόταση των εισηγητριών. Θέλω πολύ σύντομα να αναφέρω κάποια σημεία. Εγώ συμφώνησα με την προσωρινή ρύθμιση. Δεν το θεώρησα κακό να στείλουμε ένα μήνυμα δηλαδή απαγόρευσης. η οποία μπορεί να γίνει οριστική. Αλλά αν κάποια στιγμή αργότερα στο μέλλον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μπορεί να αλλάξει θέση. Έχω λοιπόν μια πιο ενδιάμεση θέση. Και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να τονίσω. Συμφωνώ με την κυρία Γιούσο. Ε, οι επιστημονικές εκθέσεις είναι πάρα πολύ εύστοχες και πάρα πολύ έγκυρες. Όταν γίνεται λόγος για δεοντολογία, ανησυχώ. Ξέρω ότι υπάρχουν διοντολογικά ζητήματα, αλλά ηθική και διοντολογία ο καθένας έχει τη δικιά του και διαλέγει κανείς όποια θέλει. Όταν ε, προβάλλουμε τέτοια επιχειρήματα σε επιστημονικές εκθέσεις ή σε δικές μας εκθέσεις, ανησυχώ, προτιμώ τις επιστημονικές. Και στις δικές μου τροπολογίες, κατανοώμεν τη δυσκολία ε, ε, εκείνων που ζητούν ε, την απαγόρευση για τα κλωνοποιημένα ζώα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως αυτό να αποδειχθεί και δεν θέλω να υπάρχουν κανόνες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεικνύονται. Κόλσον. Pan poseł Ο κύριος Νίκολσον. Οκ. Pan poseł Janusz Wojciechowski. Wojciechowski. Pani poseł Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ότι είναι απαράδεκτη η κλωνοποίηση, η απειλή για το ζώο είναι γεγονός. Και σήμερα η κλωνοποίηση ζώων είναι κάτι που μας βρίσκει αντίθετος. Αυτό είναι κοινή αίσθηση ε, και ομοφωνία. Και επίσης αντί για οδηγία θέλουμε κανονισμό και σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Ο κανονισμός ε, παρέχει το καλύτερο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και στα 28 κράτη-μέλη. Αυτό έχουμε ζητήσει και το σημαντικότερο από τη σκοπιά μας που θα πρέπει να συμπεριληφθεί είναι ότι θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιε είναι οι υπερβολικές ρυθμίσεις που μπαίνουν σε ένα τέτοιο κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το ελέγξει και να το επαληθεύσει αν υπάρχει δυνατότητα συστήματος σήμανση και να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε και το κόστος. Έτσι δεν είναι. Αν τεχνικά είναι εφικτό αυτό, δεν θα πρέπει να σημάνει επιπλέον ε, διοικητικό κόστος για τις αρμόδιες αρχές και για τους παραγωγούς και τους φορείς. Ιδιαίτερα μιλώ εδώ για τις εισαγωγές. Ε, γι' αυτό είναι σημαντικό να υιοθετηθούν και οι δικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ. Τελειώσαν εδώ οι σκιώδεις ηγητές. Ε, ένα λεπτό τώρα για τους υπολείπους. Είχαν δύο οι σκιώδεις. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ μπορούμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Φέντερλε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το πώς βλέπουμε την κοινοτομία και την τεχνολογία σε σχέση με την γεωργική παραγωγή. Πολύ συχνά υπάρχουν πολλές αυταπάτες, όμως γνωρίζουμε ότι η χρήση της κλωνοποίησης σήμερα είναι επιζήμια για τα ζώα. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστή όταν λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση και διαρκή αναθεώρηση, διότι οι τεχνικέ οι ζωοτεχνικέ μπορεί να αλλάξουν και να χρειαστεί να αναθεωρήσουμε στο μέλλον. Τι θα πει όμω διαρκή αναθεώρηση. Θα ήθελα να μου το πει και συνάδελφο από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε στην όλη συζήτηση. Είτε θα έχουμε απαγορεύσει είτε όχι και είτε θα αλλάζουμε την νομοθεσία βάσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα θέλαμε λοιπόν αναθεώρηση από την άποψη τη δική μα ομάδα να σημαίνει ότι δεν θα διατηρήσουμε εκτό. την, δεν θα αφήσουμε εκτό τις τεχνολογική εξέλιξη για τα επόμενα 20-25 χρόνια. Επίση, σημαντικό είναι οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι να έχουν ε, πρόσβαση σε υψηλή ποιότητα γενετικό υλικό για να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μουσείο ε, για το το Μουσείο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τομέα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν άλλε ήπειροι που είναι πραγματικά καινοτόμε αυτή τη στιγμή. Η κλωνοποίηση λοιπόν θα πρέπει μελλοντικά να είναι μια επιλογή εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας λόγω της, ε, της κλωνοποίησης ή των απογόνων των κλώνων και κυρίω σε σχέση με την τροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση των τροφίμων και με μεγάλη ε, προσοχή για όσα τρόφιμα προέρχονται από απογόνους κλώνων. Είναι ίσω επικίνδυνο γενετικό να τρώει κανεί κλωνοποιημένα τρόφιμα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτέ τι τεχνικέ ε, σήμερα, αλλά να είμαστε βέβαιοι για το τι είναι το γεγονό και τι όχι για την ειχνηλασιμότητα, Θα πρέπει να είναι κάτι το εφικτό, ιδίω για του απογόνους των κλωνοποιημένων ζώνων, αλλά θα επανέλθουμε στην όλη συζήτηση γιατί σίγουρα θα υπάρξουν πολλές διαφωνίες. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά τι εισηγήτριες για την έκθεσή τους. Πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ εργάστηκαν και ε, οδηγηθήκαμε σε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ανησυχώ όμω παρόλα αυτά, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι εδώ οι παρόντε, ότι η κλωνοποίηση δεν είναι προ όφελο των αγροτών. Οι καταναλωτές έχουν αντισταθεί στεναρά ε, έχουν ξεσηκωθεί απέναντι σε αυτή τη τεχνική και είναι προς το συμφέρον του ζώου, έτσι δεν είναι. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα ίδια τα κλωνοποιημένα ε, ζώα, αλλά ε, και για τους απογόνους και για τις μητέρες που εγκυμονούν και η τεχνική δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια, δεν έχει γίνει ούτε πιο φιλική προς το περιβάλλον, ούτε προ τα ζώα. Και αναρωτιέμαι αν στο μέλλον θα βελτιωθεί. Ε, και ε, ένα παραμένει ως επιλογή. Πλήρης απαγόρευση, όχι μόνο για τα ζώα ε, που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, για παραγωγή τροφίμων αλλά και για όλους τους άλλους σκοπούς. Ακούσαμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για αθλητικές διοργανώσεις που θα πρέπει να καλυφθούν. Εγώ θα το επέκτηνα και στους επιστημονικούς σκοπούς και στα κατοικίδια ζώα φυσικά να μην κλωνοποιούνται ε, για διάφορες χρήσεις. Επίσης, το θέμα αυτό της ίχνηλασιμότητας δεν μπορεί να είναι τεράστιο πρόβλημα και εφόσον υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση των καταναλωτών θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, καλυφθούν όλοι οι απόγονοι. Και αυτό πρέπει να το δούμε και στις εμπορικές συνθήκες, γιατί για λόγους εμπορικούς και μόνο γίνεται. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά που κερδίζουν. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε και το καλύτερο ε, είναι σαφέστατη σήμανση όλων των προϊόντων, όχι μόνο των ίδιων των ζώων, αλλά και των απογόνων τους. Κύριε Χόισλινγκ, ευχαριστώ πολύ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούμε στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι οι διαφορές είναι πραγματικά στις λεπτομέρειες. Και θα πρέπει να διαφωνήσω με τους φιλελευθέρους συναδέλφους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε παραθυράκια ε, του τύπου «Α, εάν γίνεται και είναι εντάξει να το επιτρέψουμε». Όχι, ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, να είναι πλήρης η απαγόρευση και όχι για να δούμε τι θα κάνουμε. Και ε, ως Ευρωπαίος αγρότης είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα γίνουμε γεωργία μουσιακού χαρακτήρα στην Ευρώπη επειδή είμαστε κατά αυτής της τεχνικής και τεχνολογίες θα πρέπει να βρούμε άλλες καινοτόμες τεχνολογίες για να προχωρήσουμε και να τις προωθήσουμε περισσότερο. Έχω ξαναπεί στη συζήτηση ότι ε, από το δίκαιο που έχουμε για την προστασία των ζώων θα πρέπει η κλωνοποίηση να απαγορεύεται από χέρι διότι προκαλεί τέτοιο πόνο και τέτοια δεινά στο ζώο που δεν χωράει καμία συζήτηση και τα τελευταία χρόνια ακριβώς δεν προόδευσε η τεχνολογία, δεν μεταξελίχθηκε ε, προς όφελος των ζώων. Παραμένει, όπως στην αρχή, είναι σχετικά ε, πολύ μεγάλα τα δεινά που υφίστανται τα ζώα. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να κοιτάξουμε και τι γίνεται με τους απογόνους. Στις εισαγωγές υπάρχει δυνατότητα να μελετήσουμε και να πούμε ε, ό,τι μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να μπορεί να ανοιχνεύεται για, με τρόπο αξιόπιστο. Στην Ευρώπη χτίσαμε ένα σύστημα μετά από πολλές αντιπαραθέσεις και, και πάθος και ε, συγκρούσεις για να ε, έχουμε μία σήμανση των ζώων και θα πρέπει να ισχύει αυτό για τα ζωικά προϊόντα, ε, για τις εισαγωγές, για τους απογόνους και θα πρέπει να το επιβάλλουμε. Και το έχουμε ξαναπεί εμείς σε μια τροπολογία και ε, επισημάναμε ότι και ο ορισμός της κλωνοποίησης δεν αρκεί, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αρκεί να περιγράψεις την τεχνική και μόνο και να το βαφτίσεις αυτό κλωνοποίηση. Γι' αυτό κάναμε και μια τροπολογία και παρακαλούμε και ελπίζουμε ότι θα τη λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο, δεν υποβάλαμε τροπολογίε. Είδαμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούσε τη σωστή κατεύθυνση, τι οποίε οι δύο συγγέτρε πολύ καλά τι συμπλήρωσαν, τι ελλείψει αυτέ. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία έχουμε σταθεί και άλλε φορέ εντάχει. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα προϊόντα που έρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, να καλύπτονται όλα τα ζώα, όχι μόνο αυτά εκτροφής ή τα είδη που αναφέρονταν στην πρώτη πρόταση. Υπάρχει το θέμα και της ε, αναθεώρησης της πρότασης κανονισμού, το πρέπει να γίνει πιο δεσμευτική και συμφωνώ με τις εισηγήτριες ότι θα πρέπει η προσωρινότητα της πρότασης αυτής να έρθει, να γίνει ε, διαρκής διότι εάν προκύψουν ε, εν καιρό ε, διαφορετικά στοιχεία για την κλωνοποίηση θα το δούμε, αλλά προ στιγμή ε, θα συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται μια δική απαγόρευση. Και όθηση από τους πολίτες και την κοινή γνώμη που έχουν δείξει την ανησυχία του για το θέμα αυτό έχουμε ήδη σημειώσει. Οπότε αυτή είναι η δική μας τοποθέτηση για το θέμα αυτό προς στιγμή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Θα δώσω 1,5 λεπτό στους ε, υπόλοιπους ε, συναδέλφου, ο κ. Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ωραία, βρισκόμαστε εκεί που έχουμε ξαναβρεθεί πριν από λίγα χρόνια. Ήμουνα κι εγώ μέλο τη ομάδα που διαπραγματεύτηκε στον τριμερή διάλογο που τελικά ναυάγησε. Είναι σαφέστατο ότι εμεί στην Ευρώπη δεν θέλουμε γάλα αποκλωνοποιημένα ζώα, ούτε κρέα αποκλωνοποιημένα ζώα και ε, κανένα στον κόσμο δεν κλωνοποιεί ζώο για να μπορέσει να το σφάξει να παράγει γάλα. Το θέμα είναι τι γίνεται με το σπέρμα και τι γίνεται με τους απογόνους. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε, διότι αυτό που είπε προηγουμένως η συγγήτρια Ρενάτε ζόμε είναι ότι δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε τελείως την εισαγωγή και να την μπλοκάρουμε από όλες τις χώρες όπου σήμερα ε, επιτρέπεται η κλωνοποίηση και διερωτώ με αν έρχεται ας πούμε μια παρτίδα κρέας από οπουδήποτε, από την Αμερική, από μια πολιτεία. Και πού θα ξέρουμε αν ο παππούς του ζώου ήταν κλωνοποιημένος ή όχι. Είναι τελείως αδύνατο αυτό. Ε, άρα θα πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστικοί, να ξέρουμε τι είναι γεγονός και τι δεν είναι. Τρεις είναι οι Είτε ε, θα απομονώσουμε ε, την δική μας την οτροφία και την παραγωγή από τον υπόλοιπο κόσμο, είτε θα αναγκάσουμε το παγκόσμιο σύμπαν να υιοθετήσει τους κανόνες μας, μπορούμε να το αποπειραθούμε, δεν ξέρω αν θα επιτύχουμε. Και το τρίτο, για τους απογόνους και τους ε, μακρινούς απογόνους, θα πρέπει να βρούμε μια ρύθμιση ρεαλιστική, εφικτή, αλλιώς συζητάμε για πράγματα που είναι τελείως ανεδαφικά ε, και πριν από τρία-τέσσερα χρόνια ήδη σπάσαμε τα μούτρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Άγνιου. Νομίζω ότι προδικάζουμε μια τεράστια παρτίδα κλωνοποιημένων προϊόντων στην αγορά και αυτό μου φαίνεται σχεδόν απίθανο. Εάν δείτε γιατί θα θέλει ένας κτηνοτρόφος να κλωνοποιήσει ένα ζώο, αυτό είναι γιατί θεωρεί ότι είναι φοβάρα υψηλής ποιότητας το ζώο του. Και θέλει όλα του τα άλλα ζώα να γίνουν ίδια. Βέβαια η φύση δεν λειτουργεί έτσι, διότι κάπου στον κόσμο κάποιο θα έχει εκτρέψει κάτι που είναι ακόμα καλύτερο και θα γίνει το δικό του κλωνοποιημένο ζώο το δεύτερο καλύτερο. Αυτό μπορεί να συμβεί. Η ακριβή παραγωγή κλώνων και τα προβλήματα που ε, προκύπτουν με την αυξημένη θνησιμότητα, σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν οικονομικά ωφέλη, για τους κλόνους τουλάχιστον. Όταν μιλάμε για απογόνους κλόνων θα πρέπει να διερωτηθεί κανείς γιατί ο απόγονος αυτός είναι κλόνος. Εφόσον ήταν μάλιστα ο άλλος, ο πρώτος, ε, το καλύτερο ζώο από όλα, γιατί να ε, ε, αλλάξει το γενετικό του υλικό με άλλα κύτταρα. Γιατί να το θέλει αυτό ένας εκτροφέας. Νομίζω ότι ανησυχούμε λοιπόν για κάτι που μάλλον δεν θα συμβεί. Αλλά ας ε, κλείσω αυτό το σχόλιο για όλους να το σκεφτούν. Ξέρουμε ότι όλοι ταξιδεύουν ε, ανά τον κόσμο πολύ γρήγορα και απροειδοποιητά μπορεί να μεταφέρουν μαζί τους και νόσους. Και υπάρχουν σε σημεία στον κόσμο όπου άλλα αγροκτήματα δεν πλήττονται από τις ζωονόσους, αλλά αλλού τα ζώα μπορεί να μολυνθούν. Σκεφτείτε λόγω χάρη την ε, αρρώστια των μελισσών πρόσφατα ε, ή ένα πρόβλημα που μπορεί να ξεκινήσει από την Ασία και να φτάσει ως την Ευρώπη, να δυσδύσει στην Ευρώπη. Με την κλωνοποίηση όμως μπορεί αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως τελικά το θετικότερο είναι να μην κάνουμε τίποτα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερχάν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς με για τον τύπο να πω ότι επιληφθήκαμε του θέματος με τρόπο πολύ περίεργο και πολύ μικρές ήταν οι προθεσμίες για ένα τόσο σημαντικό θέμα σε αυτό της κλωνοποίησης. Αυτή η ταχύτητα, αν είχε ακολουθηθεί για τους παραγωγούς ε, γαλακτοκομικών ή προκυπευτικών προϊόντων, ε, καλό θα ήταν. Η τεράστια πλειοψηφία των Ευρωπαίων, για να μην πω όλοι Ευρωπαίοι, σήμερα είναι κατά της κλωνοποίησης και των πρώτων που προέρχονται από αυτή τη διαδικασία τη είπα ισχύει το αντίθετο. Ερωτώ λοιπόν το γεγονό ότι οι διαπραγματεύσει του TTIP ζητούν κατάρριση κάποιων κανόνων ή προτύπων μας οδηγούν σε αυτή τη βεβαιασμένη συζήτηση για την κλωνοποίηση σήμερα. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κομισιόν υποκριτικά τα όσα μα λέει σήμερα θέλει από τη μία να διατηρήσει την απαγόρευση των ζώων ε, των κλωνοποιημένων, αλλά δεν είναι αντίθετα από την άλλη πλευρά στην διάθεση του εμπόριο απογόνων κλώνων ή ζώων που έρχονται από τρίτες χώρες ουσιαστικά, κλωνοποιημένων αφού αυτό απαγορεύεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κουραστήκαμε. Πραγματικά κουραστήκαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ακούμε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τελικά δεν στηρίζει σε καμία περίπτωση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ανοίγει τις πόρτες ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ε, μας αρέσει πια να μας παίρνουν για χαζούς. Βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι αρνούνται την εισαγωγή των κλώνων. Δεν αντιδρούμε όμως σωστά. Δεν πρέπει να είμαστε διαυγείς και να δράσουμε υπέρ του μέλλοντος της υπήρου μας και σύμφωνα με τις επιθυμίες των ψηφοφόρων μας. Ευχαριστώ λοιπόν τώρα η κυρία Γκροστέτ. Όπως και ο συνάδελφος Ντόρφμαν, έτσι και εγώ εκπλήσωμαι με αυτή τη συζήτηση που γίνεται γιατί εδώ και κάποια χρόνια το συζητήσαμε πιστεύω επαρκώς το θέμα. Είχαν γίνει τότε συζητήσεις περιστατωμένες, τοποθετηθήκαμε, είπαμε ότι δεν θέλουμε κλωνοποίηση και πράγματι σήμερα να για μια ακόμη φορά βιαζόμαστε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί δεν μπορώ να καταλάβω καταρχά ποιο είναι το οικονομικό όφελο. Αν ρωτήσετε του κτηνοτρόφου, ε, θα σα πω ότι δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία την κλωνοποίηση. Επομένω, ε, από αυτή τη πλευρά. Επίση, ξέρουμε ότι δεν θέλουν και οι πολίτε την κλωνοποίηση. Η ε, κλωνοποίηση ζώων είναι κόκκινο πανί. Για να μην πω πιο πολύ και από ό,τι γενικώ τροποποιημένοι οργανισμοί. Άρα, εντάξει, μπορούμε να διερωτηθούμε τελικά γιατί καλούμαστε υποχρεωτικά να το συζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποια εμπορικά ζητήματα, έχουμε το πρόβλημα των εισαγωγών. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι για την ισορροπία των εμπορικών συναλλαγών θα πρέπει και εμείς να δεχθούμε κάτι που δεν το θέλουν οι Ευρωπαίοι. Και δεν το θέλουμε στο ευρωπαϊκό έδαφος. Εγώ είμαι, όπως και η κυρία Ζόμερ, ε, ε, έχω την επιθυμία να είμαι πάρα πολύ περιοριστική και αυστηρή και σε καμία περίπτωση να θέσω ακόμα συζήτηση αυτό το οποία έχουμε ήδη αποφασίσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, το να μιλάμε για δεύτερη γενιά, για απογόνους ε, κλωνοποιημένων ζώων, χωρίς εχνηλασιμότητα, πώς μπορεί να αποδειχθεί, πώς μπορεί να είναι κανείς βέβαιος. Ε, τόσα ερωτηματικά υπάρχουν και σταματώ ε, κύριε Πρόεδρε μου, όλα αυτά τα ερωτηματικά, ε, τα ερωτηματικά αυτά τα έχουν και οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, πρέπει να τους ακούσουμε και να μην κάνουμε ό,τι να είναι. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις μόνο θέλω να κάνω. παρόλο που αν ρωτήσουμε τους ε, κτηνοτρόφους θα μας πούνε ε, ότι δεν χρειάζεται, αλλά επειδή συμβαίνει χρειάζεται ε, κάποιο πλαίσιο. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώα ε, και για τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε αθλητικές δραστηριότητες και για τα κατοικίδια και για την ειχνηλασιμότητα. όταν πρόκειται για απογόνους. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ντόρφμαν ειλικρινή απάντηση ε, μπορεί να μην ε, σας ικανοποιεί όλους, μπορεί να μην είναι καλύτερη. Δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό ε, ότι θα επιβληθεί και δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τα ίδια για κρονοποιημένα ζώα αλλά και για τους απογόνους. Μέχρι ποια γενιά παρακαλώ θέλετε να απαγορεύσετε. θα ήταν ανηλικρινές αυτό. Έχω πρόβλημα νομίζω η ειλικρινή απάντηση είναι καλύτερη, ακόμα και αν δεν ικανοποιεί τους πάντες 100%. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λουαζό. Oui, merci beaucoup. Nous devons nous opposer au clonage, bien sûr, des animaux d'élevage. Ευχαριστώ πολύ για την κλωνοποίηση των ζώων εκτροφή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από τη μια την ειχνηλασιμότητα για το κρέα, προκειμένου να προστατεύσουμε του καταναλωτέ. Και κατά τα άλλα δεν μπορούμε να ξεχνάμε και την εμπορία του ε, κρέατος, διότι καμία ειχνηλασιμότητα δεν είναι ε, βέβαιη δεν μπορούμε να ε, ανιχνεύσουμε τους ε, απογόνους των κλώνων 100%. Επίσης η κλωνοποίηση δεν έχει ε, άμεσα οικονομικά ωφέλη. Απλώς θα ετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή αγορά για την εισαγωγή κρέατος από τις ΗΠΑ στα πλαίσια της συμφωνίας TTIP και την κλωνοποίηση που ήδη, εκεί διενεργείται. ενεργείται. Επίσης θα περιορίσουμε την γεωργία με τον περιορισμό των της γενετικής ποικιλίας και ολοκληρώνοντας, επειδή θα ε, καταργήσουμε την παραδοσιακή εκτινοτροφία, που είναι και η πραγματική υπεροχή της πραγματικής γεωργίας. Να μην ξεχνάμε ότι το γεωργικό μας κεφάλαιο σήμερα προκύπτει τυχαία από τα ε, ζώα που ήδη υπήρχαν. Ε, οτιδήποτε άλλο είναι ένα αβάσιμο επιχείρημα. Ευχαριστούμε κυρία Χάγε. Ε, Ντελαή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω ότι η συζήτηση αυτή θυμίζει πολύ αυτή για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού και επίση για τα νέα τρόφιμα. Νομίζω ότι επί του θέματο θα πρέπει να διατηρήσουμε τη λογική μα και τον κοινό νου. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστέ και ρεαλιστέ και ε, θα πρέπει να βρούμε μια λύση που να είναι πιο λογική από αυτή που έχουμε βρει για τα γαματαφόμικρον όχι ευρωπαϊκή οικοδόμηση, αλλά αποδόμηση κάναμε. Ε, ευχαριστούμε ο κύριος Ντορνανό. Η κυρία Ντορνανό, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, το βρίσκω θλιβερό η συζήτηση αυτή που είναι τόσο σημαντική να είναι ευκαιρία για να διαφημίσουμε την παγκοσμιοποίηση και τις ε, ορμές της. Ε, θα πρέπει η κληροποίηση των ζώων να διέπεται από διεθνείς κανόνες. Αλλά βλέπω ότι εδώ ε, α, ουσιαστικά ομολογούμε την αδυναμία μας, την ανικανότητα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και το τι μπαίνει και βγαίνει από την Ένωση. Τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν μάλλον για κοινού κανόνες εμπορίου. Συμφωνώ με αυτό, αλλά θα έπρεπε να είμαστε υπέρ της ε, παγκόσμιας διευθέτησης. Ας προβλέψουμε ένα άλλο τροφικό ε, πρότυπο, εάν θέλουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με όλους. Ιδάλλως, Α αφήσουμε στα κάτι μέλη ε, περισσότερο δημοκρατικά ε, δημοκρατικέ οντότητε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσουν τι προτεραιότητέ του μαζί με του πολίτε του. Ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν πρόκειται να έχει καλύτερη προστασία στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσει, να εντείνει τη συζήτηση μεταξύ των κρατών προκειμένου να καταλήξει κάποιο ε, συμπέρασμα. Επίση, ε, η συζήτησή μα γίνεται εν παραλίλω με τι διαπραγματεύσει τη Συμφωνία TTIP. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προβλέψει συγκεκριμένε αυστηρέ, ε, επίσημε και μη διαπραγματεύσιμε απαιτήσει για την εκτροφή των ζώων, για τη γεωργική του εκμετάλλευση και όχι μόνο από την πλευρά τη ηθική και τη δοντολογία ή την κοινωνία, αλλά ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και την έρευνα, διότι είναι σαφέ ότι η κλωνοποίηση θα οθήσει πολλά, ε, την υποβολή πολλών γενετικών προτύπων και ε, μακροπρόθεσμα η νομοθεσία θα προβλέψει ένα σύνολο ε, γενετικών προτύπων από τα οποία δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα και δεν θα πρέπει να ανοίξουμε νέα κουτιά της Παντόρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Περίκ. Ευχαριστώ, Περί πρόκειται τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και ε, δεν είναι μόνο η κλωνοποίηση των ζώων, γιατί ε, ε, έμεσα πρόκειται και για ανθρώπους και θα πρέπει να έχουμε σαφή νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι όταν ακούτε και βλέπετε τι γίνεται εδώ, τρεις και τέσσερις γενιές σπέρμα έχουμε και ήδη πίνουμε γάλα ε, και κρέας και πού ξέρετε αν είναι κλωνοποιημένο το κρέας. Λέει ότι κανείς δεν θέλει να φάει κλωνοποιημένο κρέας. Εγώ στις Βρυξέλλες ξέρετε πόσες φορές έχω μαγειρεύσει τέτοιο κρέας ή έχω αγοράσει. Ε, εγώ είμαι κατά της κλωνοποίησης, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι ισχύει και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κάναμε μια τροπολογία, ε, συμφωνώ με την κυρία Σόμερ, για το σύστημα ίχνη λασιμότητας και για ε, για πραγματογνώμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε εδώ για αυτό το θέμα μία ώρα. Κανονικά έπρεπε να θεωρήσουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε τώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο διότι κάποιοι συνάδελφοι της ε, υπέβαλαν κάποια ερωτηματικά προς την Κομισιόν, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν για τις τροπολογίες των συναδέλφων. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στην κυρία Σαντάλ Μπουίσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ζώμα ε, που ε, παρουσίασε αυτή την έκθεση και φυσικά την κυρία Μόη. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήδη πριν από αρκετό καιρό και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2013. Και διαβάζω από τις πολλές τροπολογίες και διαβλέπω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η κλωνοποίηση ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Όλοι συμφωνούμε ότι βλάπτει τα ζώα, το είπε και η ΕΦΣ αυτό, προκαλεί πολλά δεινά στα ζώα και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος αυτή τη στιγμή ε, προσωπούν και αντιπροσωπεύουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την προτέρα κατάσταση, διότι πρώτα απ' όλα δημιουργούν νομική ασφάλεια. Θα απαγορευτεί ρητά η κλωνοποίηση, γι' αυτό είναι σαφές, ε, προς όλους τους παράγοντες και τους φορείς της αγοράς στην Ευρώπη. Τα τρόφιμα επίσης από κλωνοποιημένα ζώα θα απαγορεύονται ρητός και κάτι που έχει σημασία η απαγόρευση ε, στην πρόταση ε, ε, υπόκειται σε αναθεώρηση μετά από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά δεν είναι περιορισμένη στο χρόνο της διάρκειάς της και βάσει οποιονδήποτε επιστημονικών στοιχείων και δεδομένων που θα συλλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει αξιολόγηση. Δεν πρόκειται λοιπόν για περιορισμένη, επαναλαμβάνω χρονικά, απαγόρευση, υπόκειται σε αναθεώρηση, γιατί όλοι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ε, ε, τα επιστημονικά δεδομένα και την εξέλιξη. Η επιστήμη μπορεί να εξελίσσεται, μπορεί και να μην εξελίσσεται και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Ε, μερικά στοιχεία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας με τρόπο ρεαλιστικό και σαφή. Δεν τίθεται θέμα ευημερία των ζώων σε ό,τι αφορά ε, την αναπαραγωγή απογόνων κλωνοποιημένων ζώων. Αυτά παράγονται, αναπαράγονται με τις ε, παραδοσιακές μεθόδους. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδεχτούμε και να το αναγνωρίσουμε. Και ε, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ζώα, πρόκειται για ζώα που μπορεί να κλωνοποιηθούν, είναι πιθανό να κλωνοποιηθούν ή έχουν ζητήματα ευημερία και ευζοίας των ζώων. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά τα πτηνά ή τα ψάρια, δεν existείται τέτοιο πράγμα. Τα πουλερικά θα πρέπει να βασιζόμαστε ε, στα επιστημονικά δεδομένα, στην πραγματικότητα και σε ζητήματα ευημερίας των ζώων. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα σε σχέση με τα όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να είμαστε απολύτως συμβατοί με την αρχή της αναλογικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει και τάξει το θέμα της σήμανσης και οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας εργάζονται επί μιας μελέτης που θα εκδοθεί ε, στο τέλος του έτους για το κόστος ε, με βάση τη μελέτη αντικτύπου που κάναμε εμείς. Και θα είναι αρκετά μεγάλο σε ό,τι αφορά τη δική μας ε, γεωργία και κτηνοτροφία και ε, βιομηχανία σε περίπτωση που επιβάλλουμε σήμανση για να μην αναφέρω καν απαγόρευση ε, για τους απογόνους και τα τρόφιμα που παράγονται από τους απογόνους αυτούς. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να το στοιχειοθετεί αυτό και να συνδέεται με τις συνθήκες, ας πούμε, ε, για θέματα ευζωίας ημερίας των ζώων. Και τέλος θέλω να πω το εξής. Ο ορισμός της κλωνοποίησης ποιος είναι. Αν θέλουμε να τον τροποποιήσουμε θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι θα πρέπει να το συνδέσουμε και ε, στη μη ε, σεξουαλική αναπαραγωγή. Δηλαδή δεν είναι φυσιολογική εντό εισαγωγικών η αναπαραγωγή, έχει αναγνωρίσει η ΕΦΣΑ ότι τίθεται ζητήματα για την ευημερία των ζώων. Θα πρέπει λοιπόν οι τεχνικοί ορισμοί να ε, είναι πολύ προσεκτικοί και στη διατύπωση. Είναι ε, ειδική μορφή αναπαραγωγής αυτή. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω όλους ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί βεβαίως δεν ε, χωρών συμβιβασμό ε, στα πλαίσια του TTIP. Ε, εδώ είναι κόκκινη γραμμή αυτή. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες τις έχουμε μελετήσει προσεκτικά και φαίνεται ότι πολλές από αυτές θα σημάνουν επιπλέον μελέτη αντικτύπου. Και αυτό θα σημάνει ουσιαστικό ε, βάρος, νέα επιβάρηση και στους αγρότες κτηνοτρόφους και στην βιομηχανία. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή, μελέτη και πάντα να βασιζόμαστε στο αντίστοιχο άρθρο της συνθήκης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ τις συζήτητες πάλι. Thank you Σας ευχαριστώ για τις χρήσιμες ε, παρατηρήσεις αυτές και που μας δώσατε αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε λίγοντας, δίνοντας το λόγο ξανά στην κυρία Μόη και στην κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ όλους ε, όσοι μίλησαν. Είναι γεγονός και είναι σωστό και επανειλημμένα το είπαμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν την κλωνοποίηση. Οι πολίτες. Είναι γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αντίστοιχη ρύθμιση, μα γι' αυτό ασχολούμαστε και με το θέμα. Και επίση είναι γεγονό ότι ασχοληθήκαμε εδώ και χρόνια με αυτό το θέμα, με την κλωνοποίηση και μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε, γιατί δεν συμφωνήσαμε για ρύθμιση. Αλλά τώρα πιέζει ο χρόνο και το δείχνει και η συζήτηση που έγινε εδώ. Δεν γνωρίζουμε καν τι κυκλοφορεί ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά. Και εγώ πιστεύω ότι εκ των υστέρων ε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ό,τι κυκλοφορεί, κυκλοφορεί. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται επιγόντω να συμφωνήσουμε και να αγωνιστούμε να βρεθεί λύση. Και εγώ είμαι υπέρ μια ρύθμισης πάρα πολύ αυστηρή. Γι' αυτό ε, πρότεινα μαζί με άλλους συναδέλφου ε, να συμπεριληφθούν και ζώα που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς, καμία απολύτως εξαίρεση. Και να δούμε και για τα ε, κατοικίδια ζώα. Κάποιος το είπε αυτό. Αυτό που λέγουν στα αγγλικά pets και ζώα συντροφιάς και τέτοια. Αυτό ε, ε, το βλέπω με μεγάλη συμπάθεια, αλλά τι σχέση έχει με αυτό το κανονισμό. Δεν είναι σχετικό με το θέμα. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε, να το εντάξουμε αλλού ή κάπου σε κάποια ιδεολογική σκέψη. Γιατί στο μέλλον Όταν κάποιο του πεθαίνει και κινδυνεύει να, να πεθάνει το κανείς του, ε, το κλωνοποιούν στους δινικές για να γιατί δεν μπορούν να συνηθίσουν άλλο ζώο καινούριο, να αποχωριστούν το σκύλο τους. Ε, αυτό ε, να βρεθεί λύση δεν είναι εύκολο αλλά δεν είναι και αδύνατο. Πριν από πολλά χρόνια κάναμε τη συζήτηση αυτή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εκεί υπάρχει η και τα προϊόντα αυτά πάλι από τρίτες χώρες προέρχονται, γιατί αυτό το επιχείρημα με τις τρίτες χώρες δεν το καταλαβαίνω. Εκεί γιατί λειτουργεί η χνηλασιμότητα και δεν μπορεί να λειτουργεί στην κλωνοποίηση. Ε, και ε, δεν χρειάζεται καταρχήν ε, απαγόρευση για όλα τα ζωικά προϊόντα από χώρες όπου γίνεται κλωνοποίηση. Τώρα τίθεται το ερώτημα μέχρι ποια γενιά που ακούστηκε. Είναι γεγονό αυτό, είναι σωστό. Δηλαδή πόσες γενιές πίσω θα πάμε. Ε, θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σκεφτεί και το Συμβούλιο. Ίσως ε, αργότερα να προβληματιστούμε από κοινού. Εγώ καταρχήν πιστεύω ότι στην πράξη δεν θα τεθεί αυτό το ζήτημα γιατί δεν θα κυκλοφορήσουν τέτοια προϊόντα στην αγορά. Το ζήσαμε αυτό και με τα γενετικά τροποποιημένα. Έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις σήμανσης τώρα για ε, τρόφιμα και ζωοτροφές γενετικά τροποποιημένα, τα οποία όμως δεν κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, στα σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν δεν ανησυχώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι ως κοινοβούλιο Μπορούμε να το ζητήσουμε και για τους απογόνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο σίγουρα έχουν καταλάβει ότι εδώ είναι μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση και σίγουρα θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Γιατί θέλουν να έχουν και στο πλευρό τους το Κοινοβούλιο. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Έχω κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις και με τη συνάδελφο Τζούλια Μόιλ θα τα συζητήσω. Έχουμε και άλλα ραντεβού ορίσει για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και θα ψηφίσουμε στις 17 Ιουνίου, αν κατάλαβα καλά, θυμάμαι καλά εδώ στην Επιτροπή μας. Και αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που απομένει να κάνω είναι να υπενθυμίσω αυτό που μόλις είπατε, ότι δηλαδή η ψηφοφορία θα γίνει στις 17 Ιουνίου, στις 3 το μεσημέρι. Μαζί θα ψηφίσουμε δύο επιτροπές, να με το άρθρο 55. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο σημείο στη μέση διάταξη, οπότε μπορούμε εδώ να ολοκληρώσουμε την κοινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ τον κύριο Σικιέσκη και όλα τα μέλη των δύο επιτροπών για μια πολύ οικονομική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε 15 Ιουνίου.